Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην επαναληπτική ακρόαση του αρμόδιου για τη Γεωργία Επιτρόπου, του κύριου Βοητσεχόφσκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά που απεδέχθη τη νέα μας πρόκληση. Όπως γνωρίζετε είχαμε συνεδρίαση των συντονιστών την 1η Οκτωβρίου, αλλά δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε πλειοψηφία των δύο τρίτων, εξού και αποφασίσαμε να διαβιβάσουμε νέες γραπτές ερωτήσεις στον Επίτροπο. Όμως ε, δεν ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις γραπτές απαντήσεις που λάβαμε. Εξού και η παράκληση εκ μέρους των συντονιστών να επαναληφθεί η ακρόαση. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι έχουμε την ε, δέσμευση, ε, την προσωπική ε, ενασχόληση και ανεξαρτησία να εξασφαλίσουμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιμένουμε από όλα τα μέλη, όπως και από εσάς. Δέκα λεπτά θα σας δώσουμε για να κάνετε μια εισαγωγική παρέμβαση και θα έχετε επίσης και στο τέλος ε, της ακρόασης ένα πεντάλεπτο για μια καταληκτική παρέμβαση. Έχουμε 13 παρεμβάσεις από τους ε, συναδέλφους όπως και την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς, ε, ανά λεπτό, ε, δηλαδή ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, επερώτηση το πολύ ένα λεπτό και απάντηση επίσης για τον ψήφιπτροπο ένα λεπτό. Επτά ερωτήσεις στον πρώτο γύρο, εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και έξι ερωτήσεις ε, στο δεύτερο γύρο με βάση την κατανομή. Ε, έχουμε σε 23 γλώσσες ε, διερμηνία, μπορείτε επομένως ε, να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα όλοι και όλες, αλλά παρακαλώ να μιλάτε πολύ γρήγορα για να μπορείτε να μεταφραστείτε επαρκώς. Επίσης και στο διαδίκτυο μεταδίδεται η σημερινή ακρόαση. Επομένως, έχετε εσείς παρακαλώ τώρα κύριε υποψήφιε επίτροπε για 10 λεπτά το λόγο για την εισαγωγική σας παρέμβαση παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να γίνω σαφέστερος για το πώς θα προσεγγίσω τα καθήκοντα του Επιτρόπου Γεωργίας. Θα σας εξηγήσω πιο διεξοδικά το όραμά μου για το πώς θα καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμο, πιο φιλοπεριβαλλοντική και πώς θα καταστήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική δικαιότερη και αποτελεσματικότερη. Και τώρα θα περάσω στη μητρική μου γλώσσα, τα πολωνικά. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Οι γεωργοί είναι επιχειρηματίες και χρήζουν υποστήριξης για να, για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να τροφοδοτήσουν 500 εκατομμύρια πολίτες, να τους εξασφαλίσουν την επισητιστική ασφάλεια με υγιεινά, υψηλής ποιότητας τρόφιμα καθημερινά. Αυτό προαπαιτεί κονδύλια, χρήματα. Εγώ θα ταχθώ υπέρ ενός ισχυρού ε, επαρκούς προϋπολογισμού για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η κοινή γεωργική πολιτική προϋποθέτει και απλούστευση και εναρμόνιση. Εγώ θα υποστηρίξω και θα προτείνω τον περιορισμό της ε, επιβαρυντικής ε, γραφειοκρατίας για τους ε, γεωργούς, γιατί ο ρόλος των γεωργών είναι να καλλιεργούν τη γη και των κτηνοτρόφων να εκτρέφουν τρόφιμα. Δεν είναι δουλειά τους να συμπληρώνουν διοικητικά έγγραφα και να ασχολούνται με διοικητικέ διατυπώσει. Θα πρέπει λοιπόν να εδραιώσουμε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Γεωργία στι παγκόσμιε αγορέ. Με βάση την επιστολή ανάθεση καθηκόντων μου από την εκλεγήσα πρόεδρο Φοντερ Λάιεν, εγώ θα προωθήσω στις συνομιλίες με τους εμπορικούς μας εταίρους τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντο, του κλίματο. Τη ε, καλής διαβίωσης και μεταχείριση των ζώων, που είναι οι ψηλότερες προδιαγραφές στον κόσμο και ταυτόχρονα θα μεριμνήσω ώστε αυτά τα πρότυπα ε, και οι προδιαγραφές να τηρούνται και για τα εισαγόμενα προϊόντα, δηλαδή τις ίδιε απαιτήσει που έχουμε από τους εσωτερικούς μας, ε, από τους γεωργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τις απαιτώ και από τους παραγωγούς που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα ενισχύσω τι γεωγραφικέ ενδείξει που προωθούν και προστατεύουν την παραδοσιακή κουλτούρα τη Ευρωπαϊκή Γεωργίας. Και μάλιστα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τι χώρε τη Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κατοχυρωμένες πολλέ γεωγραφικέ ενδείξει. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, έχουμε πολλέ φιλοδοξίε σε θέματα περιβαλλοντικά και κλιματικά και θα πρέπει να τι αναβαθμίσουμε οι γεωργοί θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων, προκειμένου να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου, να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα και να υλοποιήσουμε τη μηδενική ατμοσφαιρική ρήπανση. Ήδη οι γεωργοί, καλλιεργώντας τη γη, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και υλοποιούν το ρόλο τους ε, στην προστασία του περιβάλλοντος, παρόλο που είναι τα πρώτα θύματα των κλιματικών αλλαγών, γιατί οι θεομηνίες πλήττουν και τις δικές τους καλλιέργειες και εξαφανίζουν τις οδιές του. Εγώ λοιπόν θα προστατεύσω και θα στηρίξω τους Γιώργους, όχι με προσταγές και απαγορεύσεις, αλλά με χρηματοοικονομικά ενάυσματα και κίνητρα, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι γεωργοί στην νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα προβλέψω λοιπόν κάποια οικονομικά κίνητρα για να υλοποιήσουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει οικειοθελώς να δρούν οι γεωργοί στα πλαίσια των οικολογικών προγραμμάτων και θα πρέπει να είναι ε, εθελοντικές γεωργικές δραστηριότητες υπέρ του περιβάλλοντος και στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της κοινή γεωργική πολιτικής. Εγώ θα στηρίξω και τη βιολογική γεωργία, γιατί η βιολογική γεωργία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Θα υποβάλω ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι και δίκαιη. Η γεωργία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ίδια, διαφέρει, είναι τερόκλητη και τα εργαλεία και οι μηχανισμοί της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ελαστική προσέγγιση στη χρήση των μηχανισμών και των διαφόρων μέσων. Από την άλλη πλευρά, η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να διατηρήσει αυτό τον κοινό της χαρακτήρα, τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα. Γι' αυτό εστερνίζομαι τις ανησυχίες σας που έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Χρειαζόμαστε πραγματικά μια κοινή γεωργική πολιτική που θα εδράζεται σε κοινού στόχους, σε κοινού τρόπους παρέμβασης και σε κοινού δείκτες. Και αυτό το θέμα είναι το πλέον αφιλεγόμενο στην όλη πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και είμαι απόλυτα ανοιχτός και διαλλακτικός στη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να διαφυλάξουμε τον κοινό χαρακτήρα της γεωργικής μας πολιτικής που θα μεταρρυθμίσουμε αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα διαφυλάζοντας την ευέλικτη προσέγγιση που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να βρούμε το σωστό όριο και τη σωστή ισορροπία μεταξύ της εθνικής παρέμβασης και της ανάγκης ευρωπαϊκής παρέμβασης. Η, το, ο δίκαιος χαρακτήρας της κοινή γεωρικής πολιτικής φαίνεται και στη σύγκληση, την εσωτερική και την εξωτερική. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο στην επιδίωξη της ε, εξίσωσης των ε, ενισχύσεων μεταξύ των χωρών μελών και των γεωργών στο εσωτερικό της ίδιας χώρας μέλους δεν θα πιστώ προσπαθειών προκειμένου αυτή η ευθυγράμμιση, αυτή η εξίσωση να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Γιατί η ανισότητα των ενισχύσεων είναι πολύ επώδυνο ζήτημα για πολλούς γεωργούς και κυρίως τους γεωργούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αξιότιμε προβουλευτέ, έχουμε πρόβλημα και με τη συγκέντρωση των γεών, την αρπαγή των γεών σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτά είναι θέματα αρμοδιότητας των κρατών μελών, το θέμα της κυριότητας των γεών. Αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε τους γεωργούς που απειλούνται από αυτό το φαινόμενο της αρπαγής των γεών. Οπότε, περιμένουμε ε, πολύ σημαντικές προτάσεις και η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017 περιείχε πολύ ενδιαφέρουσες συστάσεις και μέτρα. Εγώ λοιπόν θα προωθήσω τη συστάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία της αρπαγής των γεών και να προωθήσω τη την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ε, κυρίως μεταξύ των χωρών, ε, για να μιμηθούμε μάλλον τις χώρες που κατάφεραν αποτελεσματικά να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο της κερδοσκοπικής αρπαγής γεών. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία, κυρίες και κύριοι, είναι ένας χώρος στο οποίο βρίσκουν τη θέση τους διαφορετικά είδη γεωργίας. Υπάρχει χώρος και για τις μικρές και για τις μεσαίες και για τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μας εξασφαλίζουν την επισητιστική ασφάλεια. Οι μικρές όμως αγροτικές εκμεταλλεύσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη της παραμονής του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού τοπίου της υπαίθρου. Η ποικιλομορφία λοιπόν, η πολυμορφία και η ανομοιομορφία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι μια πολύτιμη αξία, είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Και αυτή την αξία και αυτό το χαρακτηριστικό στην Ευρώπη θα πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτή της πολυμορφίας. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βοτσεχόφσκι για την εισαγωγική σας αυτή παρέμβαση και θέλω να σας ευχαριστήσω που τηρήσατε και το χρόνο Θα ήθελα λοιπόν τώρα να περάσω στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και πρώτος έχει το λόγο Χέρμπερτ Ντόρφμαν εκ μέρους του ΕΛΚ. danke. Να ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριο Ριστέντα Επίτροπε. Ε, λάβαμε γραπτές απαντήσεις και διαβάζω ότι λέτε ότι τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Κομισιόνα της προηγούμενης χρονιάς της βρίσκεται σωστές σε μεγάλο βαθμό και βέβαια λέτε ότι και εσείς θα τοποθετηθεί από αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω συγκεκριμένα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες τι θέλετε να κάνετε θα ε, συνεχίσετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συμφωνήσετε με τις ε, θέσεις και θα υποστηρίξετε σε περίπτωση που χρειαστούν τριμερείς διάλογο για τις δικές μας ε, θέσεις ή θα καταθέσετε μετά τη ψηφοφορία του Κοινοβουλίου νέες προτάσεις και πώς αυτές θα σχετίζονται και με την Απράσινη Συμφωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Βοητσεχόφσκι, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν. θα σας πω το εξής. Πραγματικά ε, ζηλεύω τον ε, προηγούμενο επίτροπο, τον κύριο Τσόλος, που κατάφερε να καθοδηγήσει την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από την αρχή. Δηλαδή, είχε την πολυτέλεια να υποβάλει προτάσεις από την αρχή της μεταρρύθμισης. Εγώ ορίστηκα επίτροπος, και φαντάζομαι θα το αναγνωρίσετε, σε μια κατάσταση όπου ήδη επιτάπητος είναι έτοιμη η αναμόρφωση της ΚΑΠ. Και μάλιστα η πρόεδρος Βαντελάι με επιφόρτησε με τη διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση της ε, μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ γνωρίζω όλες τις προτάσεις Γνωρίζω και την έκθεση Dorfman που παρουσιάζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Και γνωρίζω και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου του 2019. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει αποκρισταλωθεί η θέση του τρέχοντος, της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένω φυσικά και τις νέες προτάσεις. Ένα από τα συζητήσιμα και αφιλεγόμενα θέματα είναι η διαφύλαξη του κοινού χαρακτήρα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι είμαι έτοιμος για συμβιβασμούς και είμαι διαλλακτικός ε, για να δεχτώ και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εντολή μου δεν περιλαμβάνει πρωτοβουλία δική μου για να προτείνω αλλαγές. Πάντως, οι θετικές προτάσεις που προωθούν την κοινή γεωρική πολιτική θα γίνουν δεκτές. Είμαι έτοιμος γι' αυτό. Και ήδη έχουμε τη μία και την άλλη πλευρά της συζήτησης αυτής που είναι το Συμβούλιο. Εγώ θέλω να βελτιώσουμε την κοινή γεωρική πολιτική και είμαι διαλλακτικό απέναντί σα. Είμαι πρόθυμο να εξετάσω τι προτάσει και τι δικέ σα, κύριε Ντόρφμαν, τη έκθεσή σα και την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτή η συζήτηση θα γίνει κυρίω στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου. Κύριε Ντόρφμαν, για την επερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση. Ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο, η μεταρρύθμιση αυτή ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί από 1η ε, πρώτου 2021. Επομένως, ε, πώς πιστεύετε θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή μεταβατική περίοδος. Θα πρεπει να διαμορφωθεί αυτη επαρκές διάστημα στη θέση τους οι αγρότες μέχρι να τεθεί σε ισχύ νέα κοινή γεωργική πολιτική για να προσαρμοστούν. Βοητσοχόφσκι. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της και σίγουρα θα υπάρξει και μεταβατικός κανονισμός, τουλάχιστον για την ε, πρώτη χρονιά, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της ΚΑΠ. Και η ελάχιστη διάρκεια είναι ένας χρόνος για τη μετάβαση. Εγώ, αν εγκριθώ, θα φροντίσω να διατηρηθεί αμύωτος ο ρυθμός των εργασιών και μάλιστα ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους. Οπότε, με βάση τις ε, αποφάσεις της απερχόμενης Επιτροπής, γιατί αυτό το επεξεργάστηκε η απερχόμενη Επιτροπή, ε, θα συζητηθεί και το θέμα της ε, παράτασης της τρέχουσας κάποια τουλάχιστον ένα χρόνο. Και πιστεύω ότι θα αρκέσει αυτός ο χρόνος ως μεταβατική περίοδος δεν είναι άλλωστε κάτι καινούριο. Και στις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις είχαμε μια παράταση της προηγούμενης κάπου μια μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεκάστρο έχει τώρα το λόγο. Κομισάριο. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. κύριο Ριστέντα Επίτροπε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο τομέας της γεωργίας πραγματικά απειλείται μετά από την άδεια που έδωσε ο ΠΟΕ προς τις α, αμερικανικές αρχές να επιβάλλουν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή δασμών, τιμωρητικών δασμών για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την, Αμερικανική, για την Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να δούμε τις επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα αλλά και στον τομέα της απασχόλησης από τους δασμούς αυτούς. Στην προηγούμενη σας ακροασία αναφερθήκαμε στο πώς θα καταφέρουν οι γεωργοί να επιβιώσουν στο νέο αυτό κλίμα. Συγκεκριμένα, ποια στρατηγική εσείς θα ακολουθήσετε αν αναλάβετε το αξίωμα αυτό για να αποφύγουμε μια δεινή κρίση της αγοράς που πραγματικά θα βάλει εναντίον του γεωργικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια μέτρα προβλέπονται αυτή τη στιγμή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ποια μέτρα από αυτές είστε εφαρμόστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά, κύριε υποψήφιε Επίτροπε, αν δεν καταφέρουμε δηλαδή να φτάσουμε σε μια κάποια διπλωματική λύση, την οποία όλοι προφανώς ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε. E, Σας ευχαριστώ κύριε Τεκάστρο. Ναι, ναι. Ε, γνωρίζω αυτή την κατάσταση. Ήταν πραγματικά ε, τραγική αυτή η απόφαση. Ευνηδίασε τους γεωργούς και πρώτη φορά στην ε, άσκηση παγκόσμιας ε, πολιτικής, μάλιστα εξωτερικής πολιτικής, ε, πλήττονται οι γεωργοί, που είναι τα αθώα θύματα μια σύγκρουσης και πληρώνουν τα σπασμένα αυτή της σύγκρουση. Θα μακάρι να βρεθεί μια πολιτική λύση σε αυτή τη διαμάχη που επαναλαμβάνω, δεν εμπλέκονται άμεσα οι γεωργοί. Είναι τα παράπλευρα θύματα, αθώα θύματα αυτής της κατάστασης. Μακάρι να λυθεί το συντομότερο δυνατό αυτή η διαμάχη, Αλλιώ θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό των ε, συνεπειών αυτής της απόφασης της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτές και να κινητοποιήσουμε ένα σύστημα ενισχύσεων. Στα πλαίσια της παρέμβασης αγοράς έχουμε διάφορους μηχανισμούς και εργαλεία και ευτυχώς έχουμε θετική πείρα ε, από τέτοιες καταστάσεις. Ακόμη ε, ισχύει το ρωσικό εμπάργο ο ρωσικός αποκλεισμός σε τέτοια περίπτωση που δυστυχώς συνεχίζεται αποτελεσματικά βοηθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους γεωργούς που ήταν τα θύματα αυτού του ρωσικού εμπάργου. Παρόμοιες προτάσεις θα υποβληθούν αν χρειαστεί και αν δεν διαθετηθεί προηγουμένως πολιτικά αυτή η διαμάχη. Πάντως εγώ ως Επίτροπος θα δώσω μάχη να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερα κονδύλια και να αποζημιώσουμε τους γεωργούς για τις ζημίες που ε, θα υποστούν λόγω αυτής της πραγματικά ακατανόητης απόφασης της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο κ. Δεκάστρο πάλι. Μετά την κρίση που έχουμε εξαιτία του ρωσικού αποκλεισμού, του ρωσικού εμπάρκου, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι γεωργοί μα και οι παραγωγοί μα θα συνεχίσουν να καταβάλουν το τίμημα για τι πολιτικέ επιλογέ που κάνουν τα κράτη του. Είστε έτοιμο, λοιπόν, κύριε υποψήφιε επίτροπε, να δείξετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά στο πλευρό των γεωργών και των γεωργικών επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δρομολογήσετε, θα χρησιμοποιήσετε μάλλον το απόθεμα αυτό το οποίο προβλέπετε στον κοινοτικό προπολογισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την έντονη αυτή κρίση που έχουμε στον τομέα τον παραγωγικό, το γεωργικό και στον τομέα της διανομής και πώς θα αντιμετωπίσετε με τρόπο αποτελεσματικό την έκτακτη αυτή επίγουσα κατάσταση. Εμείς θα θυμάστε ότι ως Επιτροπή Γεωργίας είχαμε ζητήσει στην επόμενη, στον επόμενο προπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής να καταφέρουμε να υπερβούμε τα 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προβλέπονται αυτή τη στιγμή. Θέλαμε να φτάσουμε στο 1,5 δισεκατομμύριο. Τι πιστεύετε εσείς κύριε υποψήφιο επίτροπε για τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση αύξηση αύξηση του προπολογισμού έκτακτη ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το απόθεμα αυτό να μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί ω αποτελεσματικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τι έντονε αυτέ διακυμάνσει που έχουμε στη γεωργική αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βοτσεχόφσκι, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για την συμπληρωματική σα ερώτηση και σα ευχαριστώ που επισημάνατε αυτό το θέμα. Θα απαντήσω σύντομα. Είμαι σαφώς υπέρ της ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων που έχουμε για να στηρίξουμε τους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης. Και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της γεωργίας. Ότι ο γεωργός κάνει τη δουλειά του και ξαφνικά ευνηδιάζεται από μια άδικη κατάσταση που εκφεύγει του ελέγχου του. Και αυτό τον οδηγεί στη χρεοκοπία, στον αφανισμό. Η εξασφάλιση λοιπόν των γεωργών έχει κέριο σημασία. Έχει κέρια σημασία. Έχουμε 400 εκατομμύρια αποθεματικό κρίση και δεν νομίζω θα είναι πιο εύκολη η κινητοποίηση αυτών των κονδυλίων γιατί υπάρχει μετάβαση από χρόνο σε χρόνο. Μακάρι να συσσωρεύονται αυτά τα κονδύλια για να αυξάνεται ο προπολογισμό του αποθεματικού κρίση. Εγώ πάντω θα υποστηρίξω οποιαδήποτε πρόταση για να βοηθήσουμε του γεωργού να εξέλθουν από την κρίση, να την αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μίλλερ. Κύριε Στέντε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που και εσείς ε, είστε υπέρ της ε, νέας ε, ΚΑΠ. Βλέπουμε και στη Γερμανία ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία για την αναδιάδρωση της εθνικής νομοθεσίας. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, αλλά χρειάζεται επίσης και προστασία του κλίματος και της βιοπικιλότητας. Είμαστε εμείς στη Γεωργία ένα τμήμα της λύσης και γι' αυτό ε, σίγουρα πρέπει να μπορούμε και να βιοποριζόμαστε από αυτή τη δραστηριότητα. Θα στοχεύσετε λοιπόν ιδιαίτερα και στους νεαρούς αγρότες. Όπως το γνωρίζετε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα ε, ότι στην Ήπεθρο ε, μόνο το 6% των είναι κάτω των 35 ετών. Κατά την άποψή σας, η μελλοντική ΚΑΠ πώς μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού ε, και τουλάχιστον στη διατήρηση του αριθμού των νεαρών αγροτών. Έχετε συγκεκριμένα μέτρα να προωθήσετε γιατί η ισχύουσα ΚΑΠ έδωσε κονδύλια ήδη ε, προς αυτό το στόχο, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Δύο Σας ευχαριστώ, κυρία Μίλλερ. Πολύ σημαντική ερώτησή σας. Φυσικά το θέμα των νεαρών αγροτών έχει κέρια σημασία για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Χρειαζόμαστε την ηλικιακή ανανέωση. Και το λέω αυτό γιατί ω μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου εκπώνησα τη σχετική έκθεση για του νεαρού αγρότε και γνωρίζω εκ του σύνεγγυ το πρόβλημα. Η έλλειψη των νεαρών γεωργών ε, είναι σημαντικό πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Γεωργία με διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα. Στη Γερμανία και στη Πολωνία, ε, μάλλον στην Πολωνία σχέση με τη Γερμανία έχουμε κάπω καλύτερη κατάσταση. Έχουμε περισσότερου νεαρού αγρότε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε αρκετά ε, ευαίσθητη, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του και να το στηρίξουμε περισσότερο. Έχουμε φυσικά τον πρώτο πυλώνα και το 2% που προβλέπεται για την αύξηση των άμεσων ενισχύσεων για τους νεαρούς αγρότες. Και έχουμε και το δεύτερο πυλώνα που, έχουμε, που προβλέπει ενισχύσεις για την πρώτη εγκατάσταση των νεαρών ε, αγροτών. Λειτουργούν αυτά τα κονδύλια, αλλά δεν αρκούν ε, αυτά τα μέσα. Γιατί είπα ε, στην πρώτη μου ακρόαση ότι έχουμε ε, όλο και λιγότερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε ένα εκατομμύριο λιγότερους ε, ε νεαρούς γεωργούς και ε, ε, οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί βιώνουν ακόμη πιο έντονα αυτό το πρόβλημα της εξαφάνισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τους νεαρούς αγρότες ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά γης. επίσης, ε, διευκολύνοντας ε, τις συνθήκες αγοράς ή περιορίζοντας την αρπαγή των γεών, πιστεύω ότι θα τους διευκολύνουμε. Είπα και στην πρώτη μου ακρόαση ότι οι γεωργοί χρειάζονται πρόσβαση στην καινοτομία, το GPS, την γεωργία ακριβίας, τα έξυπνα χωριά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσελκύσουμε με τη χρήση των τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας τους αγρότες στην Ήπεθρο, γιατί έτσι θα τους δώσουμε κίνητρα να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές. Ερώτηση συμφωνείτε μαζί μου ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες προσπάθειες ε, στο πλαίσιο της ε, κοινής πολιτική, ε, σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνιστόσα. Δεν υπάρχει διερμηνία. Δεν με ακούτε. Τώρα εντάξει, έλεγα λοιπόν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι θα πρέπει να γίνουν συλλογικέ ε, προσθέτες προσπάθειες στο πλαίσιο της κοινωνικής και της πολιτικής ό,τι αφορά την κοινωνική συνιστόσα, ε, να δοθούν κάποια σεμινάρια ανακύκλωση των γενεών, ε, κάτι το οποίο είναι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε, είναι κάτι που επιβαρύνει τους παλαιότερους αγρότες και για τους νέους αγρότες, να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και επιμόρφωση, γιατί ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πρότυπα, τα εκπαιδευτικά και τα επιμορφωτικά στην Ευρώπη ανάλογα με τη χώρα. Σίγουρα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και την καινοτομία ε, και αυτά για μένα ε, εντάσσονται στην κοινωνική συνιστόσα. Και έχετε ένα λεπτό κύριε Βουτσεχόφσκι για να απαντήσετε. Προφανώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις δράσεις για να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, ανανέωση των γενών, χάρη στη σύνδεση μεταξύ των γενών. Εγώ έχω ε, εμπειρία από την πατρίδα μου την Πολωνία. Εκεί για πολύ καιρό λειτουργήσε το σύστημα των διαθροτικών ε, επιδομάτων που έδινε κίνητρα στους πιο ηλικιωμένους ε, γεωργούς να μεταβιβάσουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, στα παιδιά τους και να εξασφαλιστεί αυτή η ηλικιακή ανανέωση. Βέβαια και η παιδαγωγική πτυχή έχει τη σημασία της, η μεταφορά τεχνογνωσίας από τους πιο ηλικιωμένους προς τους νεαρούς αγρότες. Φυσικά θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά αυτό το θέμα συνδέεται με αυτό που επισήμανε ο κύριος ε, Ντεκάστρο, την αίσθηση της ασφάλειας απέναντι στις κρίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ασφάλεια των γεωργών, να μην νιώθουν αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Γιατί υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Όσο ε, καλά και να ασκούν τις γεωργικές αρμοδιο... Ε, δραστηριότητες οι γεωργοί, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χάσουν τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την αίσθηση της ασφάλειας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για να προσελκύσουμε και νεαρούς αγρότε να ασχοληθούν με τη γεωργία. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε. Είναι πολύ πιο ε, μέχρι τώρα συγκεκριμένες απαντήσεις από το πρώτο γύρο της ακρόασης. Αυτό είναι θετικό και αυτό που είπατε για την οικολογική γεωργία. Θέλετε ένα σχέδιο δράσης, ε, θέλετε συγκεκριμένα πρότυπα, αλλά θέλετε επίσης να αγωνιστείτε και για την ε, εξωτερική μετατροπή και σύγκληση. δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα. Εσείς θα ε, εστιάσετε στο να δοθούν περισσότερα χρήματα στις μικρότερες και λιγότερες μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, έχουμε το 40% αυτών των ε, μέτρων. Πιστεύουμε όμως ε, ότι θα είναι πιο μεγάλες επιπτώσεις από αυτές που εσείς επιθυμείτε σε ό,τι αφορά τη δεσμευτικότητα. τι θα κάνετε για τη δεσμευτικότητα των μέτρων και αν θα περιληφθεί η ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών ε, στα μέτρα επιτήρησης και πώς ε, την επανεθνικοποίηση της κοινής πολιτικής θα την αποφύγετε για το Μερικοσούρ. Ένα τελευταίο σημείο. Υπάρχουν αυτές οι προτάσεις επιδοτήσεων των ψυχανθών μεταξύ άλλων. Τι θα κάνετε εσείς και τι θα δώσετε ως οδηγές στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ε, αναφέρθηκα εκτενώς στο θέμα αυτό στην πρώτη μου ακρόαση. Φυσικά είμαι υπέρ της προστασίας των μικρών εκμεταλλεύσεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ευνοιοκρατία υπέρ των μικρών εκμεταλλεύσεων. Όχι, δεν τις ευνοώ. Απλώς ε, εκ των πραγμάτων είναι πιο αδύναμες οι μικρές εκμεταλλεύσεις και πιο ε, ευάλωτες. Γι' αυτό θέλουμε να τις προστατεύσουμε και στα εθνικά στρατηγικά σχέδια ελπίζω να υπάρχουν και οι μηχανισμοί προστασίας των μικρών εκμεταλλεύσεων ώστε να μην χάσουμε τους μικροκαλλιεργητές, να μην εξασφανιστούν από το ευρωπαϊκό τοπίο. Γιατί ε, αν δεν διατηρηθεί η ποικιλομορφία τη ευρωπαϊκή Γεωργία, θα οδηγούμε το αυτοκίνητο στην Ευρώπη και θα νομίζουμε ότι είμαστε στον Καναδά με μεγάλε μόνο εκμεταλλεύσεις. Φυσικά θα πρέπει να διαφυλάξουμε το γεωργικό μα μοντέλο που όπω σα είπα είναι ανομοιόμορφο και αποτελείται από διάφορε μορφέ εκμεταλλεύσεων μεγάλε και μικρέ. Σε ό,τι αφορά τι πρωτεϊνούχε καλλιέργειε και τα ψυχανθή, είμαστε μεγάλη εισαγωγή σόγια από την Αμερική. 36 ε, και εκατομμύρια τόνοι το χρόνο είναι οι εισαγωγέ μα σόγια. Και μακάρι ένα μεγάλο τμήμα αυτών των εισαγωγών να το αντικαταστήσουμε από τοπική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα με κλειστό ε, κύκλο παραγωγής, με την παραγωγή στο αγρόκτημα των ζωοτροφών για την εκτροφή των ζώων και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλά κονδύλια που προβλέπονται στο δεύτερο πυλώνα, Οπότε έτσι μπορούμε να μειώσουμε και τις αγωγές, να μειώσουμε τις ε, μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις, να στηρίξουμε την καλή διαβίωση και καλή μεταχείριση των ζώων και να στηρίξουμε ταυτόχρονα τις μικρές καλλιέργειες με ένα τέτοιο πρόβλημα, πρόγραμμα κλειστής ε, ή βραχαίως κυκλώματος ε, παραγωγής. Εγώ θα φροντίσω και θα προτείνω τη συμπερίληψη τέτοιων μηχανισμών στα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Έχετε ένα λεπτό για την υπερώτησή σας. Σε ό,τι αφορά τη σημευτικότητα και τα μέτρα κλιματικής αλλαγής θα φροντίσετε να τηρούνται ομοιόμορφα αυτά και να μην υπάρχουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, αν θέλετε να ενισχύσετε πολλά μέτρα για το δεύτερο πυλώνα, θα πρέπει και εσείς ε, να τα υποστηρίξετε αυτά ως Επίτροπος. Δηλαδή, οικονομικά αυτός ε, ο πυλώνας ο δεύτερος να μην, ε, να μην έχει ως το 30%. Τι θα κάνετε λοιπόν, θα ενισχύσετε ή θα θα βοηθήσετε να μην αποδυναμωθεί η προκοδότηση του δεύτερου πυλώνα. Ένα λεπτό έχετε κύριε Βολτσιαχόφσκι. Η ερώτηση για τον προπολογισμό, η ενίσχυση του πρώτου ή του δεύτερου πυλώνα με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί μακάρι να είχαμε πιο γενναιόδωρο γεωργικό προϋπολογισμό. Θα ήμουν πανευτυχής αν ε, ο γεωργικός προϋπολογισμός παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα. Και ακόμη πιο ευτυχής θα ήμουν αν αυξανόταν κιόλα. Θα ήταν τεράστια ευτυχία για μένα να έχουμε δαψιλή γεωργικό προϋπολογισμό για να τον κατανείμουμε δίκαια στους Ευρωπαίους γεωργούς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο προϋπολογισμός έχει το επίπεδο που έχει. Και σίγουρα θα βρούμε ε, επιχειρήματα για έναν ισχυρότερο γεωργικό προϋπολογισμό. Εγώ θα ταχθώ υπέρ ενός επαρκούς προϋπολογισμού για τη γεωργία και θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει υπό χέρι μου, ώστε ο γεωργικός προπολογισμό να ανταποκρίνεται στις, προ... στις προσδοκίες των Ευρωπαίων γεωργών. Δυστυχώς όμως πέρασε το λεπτό που είχα για την απάντηση στην επερώτησή σας. Ευχαριστώ κύριος Νταβίδ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Στην εισαγωγική σας παρέμβαση αναφερθήκατε σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα και ήδη πολλές ερωτήσεις ετέθησαν από τους συναδέλφους, τις οποίες ήθελα να θέσω κι εγώ. Πάντως, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα στο οποίο θα περίμενα να δώσετε μια σαφέστατη απάντηση. πώς μπορούμε να ευνοήσουμε περισσότερο εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα από την Ουκρανία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τις χώρες του Μερκοσούρ, Βιετνάμ, Ηνωμένε Πολιτείε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τις εισαγωγέ αυτές. Αποδέχεστε εσεί τον ανταγωνισμό αυτό που έχουμε από τα γεωργικά αυτά προϊόντα, ο οποίο θεωρώ ότι σε ορισμένε περιπτώσει είναι σαφώ αθέμητο και δυστυχώ πολλέ φορέ οδηγεί σε μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, πολλές φορές σε αδυναμία των γεωργών να ανταπεξέλθουν απέναντι στον θέμητο αυτό ανταγωνισμό. Τι προβλέπετε εσείς να κάνετε σε σχέση με αυτό. Δύο λεπτά κύριε Βοτσεχόφσκι για την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταβίτ, κύριε Ευρωβουλευτά για την ερώτησή σας. Ναι, φυσικά πρέπει να προσπίσουμε το εισόδημα των Ευρωπαίων Γεωργών απέναντι σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Απ' την άλλη, χρειαζόμαστε και το διεθνές εμπόριο. Από πολλές απόψεις, οι εμπορικές συμφωνίες είναι ευνοϊκές για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την Ευρωπαϊκή Γεωργία πολλές φορές, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εξαγωγέας ε, τροφίμων. Έχουμε πλεόνασμα στις, εμπορικές, στη, στις εξαγωγές μας στα τρόφιμα. Οπότε είναι χρήσιμες οι εμπορικές συμφωνίες, αλλά δεν θα πρέπει τα κέρδη για ένα κλάδο να γίνονται εις βάρος ή να αποκομίζονται εις βάρος ε, ή στην πλάτη άλλου κλάδου. Δεν θα πρέπει οι γεωργοί να είναι τα θύματα στο βωμό των εμπορικών συμφωνιών. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους γεωργούς. Βέβαια θα πρέπει μόνο μερικοί γεωργοί να ε, έχουν κέρδη από τις εμπορικές συμφωνίες και άλλοι μόνο ζημίες. Επαναλαμβάνω, ως Επίτροπος Γεωργίας θα δώσω μάχη για να προστατεύσουμε τους ε, γεωργούς σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Και θα πρέπει η οι δασμολογικέ ποσοστώσεις για τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ευρώπη να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απειλούν τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Βέβαια, σε ακραίε περιπτώσεις και αν έχουμε όντω ζημία των γεωργών, θα κινητοποιήσω βοηθητικά εργαλεία, τους μηχανισμούς που έχουμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων που υπάρχουν, μας το υπενθύμισε και ο κύριος Δεκάστρο, και όπω είπε και εκείνο, θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα αποθεματικά τη κρίση, αυτού του μηχανισμού αντιμετώπιση των κρίσεων, για να μπορούμε αποτελεσματικά να αντιδρούμε σε περίπτωση κρίση. Ερώτηση του κύριου Ντάβιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο δίκαιη κατανομή των γεωργικών επιδομάτων και ενισχύσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ισχύουν διαφορετικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες από ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε για τις διαφορές αυτές. Δεν θα πρέπει να επιδείξουμε απλώς γραφειοκρατική αδιαφορία, έτσι δεν είναι. Ε... Σας ευχαριστώ. Μίλησα προηγουμένως για την εσωτερική και εξωτερική σύγκληση που απαιτείται. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εξισώσουμε τις ενισχύσεις μεταξύ των γεωργών και των γεωργών ε, σε διαφορετικές χώρες αλλά και των γεωργών εντός της ίδιας χώρας. Μερικές φορές είναι ένα προς δέκα οι διαφορές. Υπάρχουν γεωργοί που λαμβάνουν δεκαπλάσεις ενισχύσεις από άλλους. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις ε, διαφορές να τις εξορροπήσουμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για την επίτευξη της εσωτερικής και της εξωτερικής σύγκλησης. Και ήδη είμαστε στο σωστό δρόμο για να μειώσουμε αυτές τις διαφορές και στο μέλλον να τις, εξ, να τις εξορροπήσουμε πλήρως. Πάντως, έχουμε ανάγκη μια περισσότερο φιλόδοξη πολιτική και πιο α, σημαντικές αποφάσεις. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη πυγμή και αποφασιστικότητα γιατί αυτό το θέμα των άνισων ενισχύσεων πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες και να υλοποιήσουμε αυτή την εξορόπιση των ενισχύσεων, την σύγκληση δηλαδή. Ο κύριος Κουσμιούκ, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ε, αναφερθήκατε ήδη στο θέμα της συγκέντρωσης των ε, ευρωπαϊκών γεωργικών γεών η κυρία Νόιχλ εκπώνησε σχετική έκθεση που μάλιστα εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σημαντική πλειοψηφία. Και φαίνεται από την έκθεση αυτή το 2013 το 3% ε, των ε, γεωρικών ε, εκμεταλλεύσεων έλεγχε το 50% των γεών και 76% ε, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έλεγχαν το 12% των γεών. Οπότε υπάρχει μεγάλος ε, ανταγωνισμός και αθέμητος ανταγωνισμός. Πάντως μερικές χώρες όπως η Πολωνία ε, έχουν ήδη αποτελεσματικά καταπολεμήσει αυτή τη συγκέντρωση γεών. Θα πρέπει όμω να χρησιμοποιήσουμε και κάποιου μηχανισμού τη κοινή γεωργικής πολιτική για να αποτρέψουμε αυτή τη συγκέντρωση των γεωργικών γεών και η ευρωπαϊκή γεωργία, το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας να στηρίζεται κυρίω σε οικογένειακέ αγροτικέ εκμεταλλεύσεις. Βοητσεχόφσκι, σα ευχαριστώ. Γνωρίζω την έκθεση τη κυρία Νόιχλ για το θέμα αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά συνταρακτικά αυτά τα αποτελέσματα ε, τόσο σημαντικής συγκέντρωσης των γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ε, ανησυχητική η κατάσταση και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Φυσικά δεν θα πρέπει να σφετεριστούμε τις εθνικές αρμοδιότητες, γιατί με βάση ε, το άρθρο 345 της ηθικής για τη, λειτουργία, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα κυριότητας, ιδιοκτησίας των γεών είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη διατάξεις για το ποιος δικαιούται να αγοράζει γέες αγροτεμάχια και να ε, ασχολείται με τη γεωργία. Πάντως μπορούμε να περιορίσουμε τις ε, υπερβολικέ συγκεντρώσεις, χωρί να παραβιάζουμε τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επίσης, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τις διακρίσεις. Δεν μπορεί μια χώρα να θεσπίζει διατάξεις που να περιορίζουν τους ε, υπηκόους άλλων χωρών να αγοράζουν ε, γεωργικές γέες. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τις διακρίσεις, να προωθήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γιατί αναφέρατε το πολωνικό παράδειγμα. Γνωρίζω την σχετική νομοθεσία και όντως χάρη στις νομοθετικές αυτές διατάξεις καταπολεμούμε την υπερβολική συγκέντρωση των γεωργικών γεών. Η Πολωνία θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, αλλά και άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της συγκέντρωσης των γεών και να προστατεύσουμε τους γεωργούς από την αρπαγή των γεών. Ένα μηχανισμός θα ήταν ίσως ε, το κάπινγκ, η εφαρμογή ανωτά του ορίου ε, σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις για τις ε, μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το ανώτατο όριο να είναι τα 100.000 ευρώ. Και αυτό το θέμα όμως είναι από τα πιο συζητήσιμα και αφιλεγόμενα των προτάσεων μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο κύριος Κούσμιου για επερώτηση. Θα συνεχίσω στο ίδιο θέμα. Μήπως θα πρέπει να προσδιορίσουμε την έννοια του ενεργού γεωργού για να αποφύγουμε τις έμεσες ενισχύσεις ε, της ΚΑΠ ε, σε γεωργούς που δεν είναι πραγματικά γεωργοί κατά κύρια απασχόληση γεωργοί και έτσι εμέσως να περιορίσουμε και τη συγκέντρωση των γεωργικών γεών. Συμφωνώ μαζί σας ότι όντως αυτό θα ήταν ένα σημαντικός μηχανισμός για να περιορίσουμε την εκμετάλλευση της κοινή γεωρικής πολιτικής από κάποιους που δεν είναι γεωργοί. Γιατί η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να προορίζεται για τους πραγματικούς γεωργούς. Και έχουμε στα πλαίσια του ορισμού του ενεργού αγρότη ε, κάποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν φυσικά και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το ρόλο τους. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι είμαι διαλλακτικός και ανοιχτός. Αν υπάρξει πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι πρόθυμος να την εξετάσω. Αλλά φυσικά θα πρέπει να λάβω υπόψη και τη θέση του Συμβουλίου. Η πλειοψηφία του είναι κατά του κοινοτικού ορισμού του πραγματικού αγρότη. Πάντως, ε, αυτά τα 365 δις που προβλέπονται στο κοινοτικό προϋπολογισμό ε, μακάρι να αυξηθούν και αυτά τα κονδύλια να προορίζονται για τους πραγματικούς, για τους γνήσιους γεωργούς, για τους ανθρώπους δηλαδή που ασχολούνται κατά κύρια απασχόληση με την ε, γεωργική δραστηριότητα. Κύριο κύριος Φλάναγκαν. ευχαριστώ πολύ που είστε πάλι παρόν εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάτε επίση στην ε, μητρική σα γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε τη μητρική μα γλώσσα, διαφορετικά τη χάνουμε. Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά στην Ιρλανδία. Πρέπει να σας πω ότι έχετε δημιουργήσει αρκετές συνθήκες ελπίδας και αισιοδοξία, θα έλεγα, ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές. Προέρχεστε όμως από την ίδια πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν και οι συντηρητικοί του Ηνωμένου Βασιλείου που θυμάστε ότι κάνανε κάποιες δηλώσεις για την Πράσινη Συμφωνία χωρίς όμως να δώσουν επί τα συνέχεια. Νομίζω ότι στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική έχετε τα 20 teams, τα οικολογικά συστήματα. Προβλέπετε ένα 20%, ένα 30% έχει ζητήσει η Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ποια είναι η δική σα η τοποθέτηση, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, ιδίω στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Εμεί έχουμε αποκρισταλώσει τη δική μα τη θέση. Περιμένουμε τη δική σα την τοποθέτηση. E, e, Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε και από την προηγούμενη ακρόαση, είμαι υπέρ της κοινή γεωρικής πολιτικής που θα είναι ταυτόχρονα και περιβαλλοντική. Και μάλιστα η προτινόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, είναι λογική σε κάποιο βαθμό είναι υποχωρεωτική, προβλέπει κάποια αιρεσιμότητα για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά ταυτόχρονα έχει και θελοντικά οικολογικά συστήματα και προγράμματα και προαιρετικέ δράσει στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Και το 20% που αναφέρεται ε, στην Επιτροπή Γεωργία είναι καλό σημείο αφετηρία και είμαι ανοιχτό για να το συζητήσουμε περαιτέρω πριν ε, αρχίσουμε να μιλάμε για συμβαστικές λύσεις, θα πρέπει πρώτα να δούμε όλα τα, όλες τις προτάσεις που έχουμε επιτάπητος. Και ας μην ξεχνούμε και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Πάντως, αν μου δώσετε την έγκρισή σας και αναλάβω σε επίτροπος, θα συζητήσω για τα θέματα αυτά με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Το 20% είναι μια λογική πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της πρότασης και θα την υποστηρίξω. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα ή χρειάζεται υψηλότερο ποσοστό, ας δούμε και τη θέση των υπόλοιπων ενδιαφερομένων και των άλλων πλευρών και κυρίως τη θέση του Συμβουλίου. Τώρα, για την προστασία των ζώων. Σίγουρα το θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Αλλά δεν ε, θα αναλάβω πρωτοβουλία για επιβολή περαιτέρω απαγορεύσεων σε σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα. Γιατί ήδη έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υψηλότερες παγκοσμίες προδιαγραφές για την ευζοία, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Εγώ α, θα ταχθώ υπέρ της προαιρετικής αναβάθμισης από πλευρά κτηνοτρόφων των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων. Ευχαριστώ. Καλαβαίνω απόλυτα για ποιο λόγο θέλετε να προωθήσετε μια εθελοντική προσέγγιση από πολιτική πλευρά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα είναι εθελοντικό για ορισμένου και όχι για άλλου τελικά. Και τελικά αυτό που θα δούμε είναι ότι στι πιο δύσκολε περιοχέ να υπάρχουν γεωργοί οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τελικά όλο το άγχο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Πάντω, ε, Ποια είναι η δική σας η άποψη όσον αφορά τα 20, 20 schemes θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένε ενισχύσει για συγκεκριμένε γεωργικέ υπηρεσίε, γιατί στην Ιρλανδία αλλά και σε άλλε χώρε βλέπουμε την εξή κατάσταση. Με έναν κάπω μαγικό τρόπο φυτεύουμε δέντρα τα οποία απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα χρηματοδοτικό κίνητρο γι' αυτό προβλέπεται με ένα τέτοιο κίνητρο, για παράδειγμα, όσον αφορά την δέσμευση και απορρόφηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να απορριθούμε όλο περισσότερο όσον από συγκεκριμένε πρακτικέ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένε τέτοια κίνητρα. Υπάρχουν για του τυρφώνε, για παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ανάλογα παραδείγματα κι αλλού. Ευχαριστώ. Αυτά τα ζητήματα που επισημάνατε είναι από τα πιο εμφυλεγόμενα. Τα οικολογικά προγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται κυρίως από τα κράτη-μέλη. Αλλά θα έχουμε και κάποια ευρωπαϊκά οικολογικά προγράμματα που είναι μέσα στον κατάλογο των, το κατάλογο δραστηριοτήτων μας. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Εγώ είμαι υπέρ να έχουμε και κάποια οικολογικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Προβλέπονται ήδη ε, για τους τυρφώνες, για κάποιες ε, ζώνες οικολογικής εστίασης και η ζώνη των 10 μέτρων ε, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βιοπικιλότητα οι, βοσκο, οι βοσκότοποι, οι μόνιμοι και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τέτοια μέτρα οικολογικά. Μακάρι να υπήρχαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μην αφήσουμε στη μοίρα τους τα κράτη-μέλη και να είναι μόνο αυτά επιφορτισμένα για την υποβολή τέτοιων προγραμμάτων οικολογικών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων, οπότε προχωρούμε τώρα σε άλλους ερωτώντες με πρώτη κυρία Σμιτ Μπάουερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Οριστέντα Επίτροπε πολλά κράτη-μέλη προχωρούν ε, στη χάραξη αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα ε, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την άνθηση της υπέδρου των αγροτικών περιοχών. Το έχουν αναφέρει το θέμα αυτό οι προλαλήσαντες. Πραγματικά υπάρχουν ε, πολλές περικοπές στον προϋπολογισμό και ήδη και στην προηγούμενη σας ακρόαση αλλά και τώρα μιλήσατε για την ανάγκη να υποστηριχθούν οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ότι χρήζουν υποστήριξη. Αλλά θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Μιλήσατε για το σχέδιο δράση. Για μένα, ένα παράδειγμα ε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και μην ξεχάσετε, ε, όταν μιλάτε για του μικρού αγρότε και για τι αγροτικέ μεταλλεύσει, να μιλάτε και για τα εσωρινέ και τι ε, λιγότερο ανεπτυγμένε, τι υποβαθμισμένε περιοχέ που και εκεί πρέπει να στηρίξουμε την υπεθρο. Υπάρχουν πολλοί οποίοι φεύγουν. Έχουμε την απερίμωση των περιοχών αυτών δεν είναι κατάλληλες ε, και οι υποδομές ή στη συνέχεια και οι υποδομές φθήνουν λόγω της ε, εγκατάλειψης αυτών των περιοχών. Έχετε δύο λεπτά κύριε Βουτσίεχοφσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Και εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για την αγροτική ανάπτυξη είναι χαμηλότερος από ό,τι στην, περίοδο, στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Γιατί προβλέπεται αύξηση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης. Για να ε, κρατηθεί αυτό το κονδύλιο στα προηγούμενα επίπεδα θα πρέπει να αυξηθεί το, η εθνική συνεισφορά. Και σίγουρα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απερίμωση της υπαίθρου. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη. Και στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μας ε, για την ε, χρησιμοποίηση των κονδυλίων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην γίνεται κακή χρήση των κονδυλίων, να πιάνουν τόπο, να φτάνουν πραγματικά στους δικαιούχους που πραγματικά χρειάζονται τα κονδύλια για να εξυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Αλλά δεν θα πρέπει τα περισσότερα κονδύλια να αφιερωθούν σε αυτό το θέμα του εξυγχρονισμού, παρόλο που είναι απαραίτητο θα πρέπει τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να παραμείνει ο πληθυσμό στην ύπεθρο, στι αγροτικέ περιοχέ και στις ορεινέ περιοχές και στις πιο απομακρυσμένες. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τον αφανισμό της γεωργίας σε αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να παραμείνουν και στις ορεινές περιοχές οι γεωργοί και να τους στηρίξουμε περισσότερο από την κοινή γεωργική πολιτική. Και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να προωθήσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγωγών και των τοπικών ε, μεταποιητών. Γιατί αν στηρίξουμε τη βιολογική γεωργία και αν έχουμε ειδικέ προϋποθέσεις ε, για τις εκτροφές, να στηρίξουμε και την τοπική γεωργία και κτηνοτροφία. Οπότε αν οι βιομηχανίες μιας συγκεκριμένης περιοχής ή μεταπίτες αγοράζουν τοπικά, θα ενισχύσουμε έτσι έμεσα και την τοπική καλλιέργεια. Η κυρία Φοντελάν έκανε κάποιες προτάσεις ε, για το κλίμα, το περιβάλλον ε, και είπε ότι θα πρέπει και ε, η Γεωργία να βοηθήσει με περικοπές, παραδείγματο χάρη, στο πλαίσιο της νέας κοινωνικής πολιτικής. Πώς μπορεί με λιγότερα κονδύλια να προστατευτεί καλύτερα το κλίμα και εμείς οι βουλευτές από την Επιτροπή Γεωργίας χρειαζόμαστε έναν ισχυρό εταίρο στο πλευρό μας για την επόμενη πεντέτεια. Θέλουμε το ξέρουμε αυτό και ξέρω, εσείς ως ε, οριστής επίτροπος, είστε ο δικό μας επίτροπος, είστε αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί στο πλευρό μας ε, και αν χρειαστεί κιόλα ε, να αντιπαραταχθείτε στο σώμα των επιτρόπων για μια βιώσιμη γεωργία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Σμιτμπάουερ. Φυσικά θα ήθελα να κάνω αυτή τη δήλωση. Είμαι έτοιμος για μάχη. Ε, είμαι έτοιμος ακόμη και να αντιπαραταχθώ ε, στους άλλους επιτρόπους. Και όποιος ε, ισχυριστεί ότι δεν χρειάζονται χρήματα οι Ευρωπαίοι Γεωργοί ή θα πρέπει να περικοπούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, θα με βρει απέναντι. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι χρήζουν τεράστια υποστήριξη, γιατί η κατάσταση είναι δεινή πραγματικά για αυτού. Θα πρέπει να του προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε του αγρότε μα. Και δεν είναι τυχαίο που σα είπα ότι καθημερινά χάνουμε χίλιε αγροτικέ εκμεταλλεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαφανίζονται, αφανίζονται, χρεοκοπούν χίλιε εκμεταλλεύσει καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον, ε, στο επόμενο ΠΔΠ και θα δώσω επιχειρήματα ε, που να συνηγορούν υπέρ της ενίσχυσης της υποστήριξης των Ευρωπαίων Γεωργών και Κτηνοτρόφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο συνάδελφος κύριος Ολέκας. Σας ευχαριστώ, κύριε υποψήφιε επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ακούσαμε σήμερα πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις μας και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Αναφερθήκατε όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στην ακροτική ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ γι' αυτό διότι η ζωή στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει, αν θέλετε, συγκεκριμένες επιλογές ζωής. Επομένως, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με συγκεκριμένε δράσει που θα μπορούσατε να αναλάβετε προκειμένου να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και να υπάρχουν καλύτερε υποδομέ στις αγροτικέ περιοχέ, βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και το ζήτημα τη σύγκληση επίση. Πώ μπορεί να εφαρμοστεί και αυτό στις αγροτικέ περιοχέ, Θα μπορούσατε να μα δώσετε πιο συγκεκριμένε απαντήσει όσον αφορά τη σύγκληση. Αναφερθήκατε κυρίω στην εσωτερική σύγκληση και ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και αποκλήσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η δική σα λοιπόν η θέληση, η θέση όσον αφορά τις ενισχύσεις. Μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον μέσες ενισχύσεις κοινέ για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Zrobię wszystko, co możliwe, żeby... E, Θα φροντίσουμε ώστε να εξισώσουμε τις άμεσες ενισχύσεις το συντομότερο δυνατό, να επιτύχουμε αυτή την σύγκληση. Το είπα και στην ε, προφορική μου δήλωση. Βέβαια αυτό δεν ε, ε, επαφίεται μόνο σε έναν επίτροπο. Θα πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση για να υλοποιήσουμε αυτή τη σύγκληση. Πάντως, ήδη έχουμε συμφωνήσει ότι υπάρχει ανισορροπία και ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι άδικο και δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Το 2004 ε, είχαμε την ε, μεγάλη διαβρύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει σχεδόν 16 χρόνια από την ε, ένταξη αυτή. Δεν θα πρέπει να εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το χάσμα μεταξύ παλιών και νέων ευρωπαϊκών χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να υλοποιηθεί αυτή η ευθυγράμμιση των ενισχύσεων. Και φυσικά η σύγκληση δεν θα πρέπει να πλήξει τους γεωργούς των παλιότερων χωρών, θα πρέπει να βρούμε δίκαιες λύσεις για όλους και είμαστε σε καλό δρόμο. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, αυτό που ρωτήσατε κύριε Ολέκας, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν το ανέφερα ακόμη, αλλά θα πρέπει να το πούμε. Το θέμα της ε, υποστήριξη της υπαίθρου και από το Ταμείο συνοχή και από τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Γιατί δεν έχουμε μόνο για την ανάπτυξη της αγροτικής, των αγροτικών περιφερειών μόνο το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς για να βελτιώσουν τις βιωτικές τους συνθήκες στην Ήπεθρο. Και γι' αυτό θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε περισσότερο και από την πολιτική συνοχή και όχι μόνο από τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό θα επιχειρήσω. Η επερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την απάντηση που μόλις δώσατε. Νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι συγκλίνουν οι απόψεις μας. Ωστόσο, Ξέρετε ότι είμαστε σε χώρες ε, οι οποίες έχουν ένα σοβιετικό παρελθόν και θυμάστε το αστείο αυτό, το οποίο να πάρα πολύ, ότι οι κομμουνιστές μας είχαν ε, υποσχεθεί ένα πολύ πιο φωτεινό και λαμπρό μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στο εγγύ μέλλον να κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πρόσβαση σε μία τουλάχιστον μέση τιμή όσον αφορά ε, τι γεωργικέ ενισχύσει. Ευχαριστώ. Κύριε Βουτσεχόφσκι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά θα το προσπαθήσω, τουλάχιστον στη διάρκεια της θητείας, να το πετύχω. Πολύ σύντομη. Πολύ σύντομη απάντησή σα. Ε, σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσιόλος. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Βλέπω ότι αυτή τη φορά, στη δεύτερη σα αυτή ακρόαση, είστε πολύ πιο συγκεκριμένο στι απαντήσει που δίνετε και ακριβώ αυτό θέλουμε και εμεί, διότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να αποτελεί πρωτερχική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ξεκινήσουμε από τη βασική ιδέα ότι η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να ασχοληθεί και με την πτυχή των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων γιατί αυτό ζητούν άλλωστε και οι πολίτες, αλλά θα πρέπει επίσης ε, να συμβάλλει στην ε, κλιματική αλλαγή, στην αντιμετώπιση μάλλον της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να προωθεί συγκεκριμένε ε, φύλλο-περιβαλλοντικές πολιτικές εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο για τους γεωργούς. Θα ήθελα να γνωρίζω δεδομένων όλων αυτών πώς μπορεί να κινηθεί η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής προκειμένου να μπορούν να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι παράλληλοι στόχοι. Και επίση, να δούμε επίση πώς θα καταφέρουμε να, να εφαρμόσουμε του φιλοπεριβαλλοντικούς μηχανισμούς. Ξέρετε ότι ε, για το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος προβλέπεται στο τμήμα του κοινοτικού προπολογισμού συγκεκριμένη ποσοστά. Εσείς ποια ποσοστά θέλετε για τα ecosystems, για τα οικολογικά αυτά συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιόλος. Κύριε Επίτροπε θα έπρεπε να πω δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, η κυρία Φοντερλάιν μου ανέθεσε μεταξύ άλλων ε, και το καθήκον ε, του να αναπτύξω ένα όραμα για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου των αγροτικών περιοχών. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις, ε, πόσο ποσοστό εξ αυτών είναι μικρές επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να το κάνουμε από κοινού, μαζί με το Κοινοβούλιο, μαζί και με τους αγρότες και ε, τις διάφορες ενώσεις ε, και θα το προσπαθήσω και εγώ στο πλαίσιο της θητείας μου. Για αυτά τα οικολογικά εργαλεία που έχουμε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η, η συμπερίληψη της Γεωργίας σε αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ένταξη της Γεωργίας σε αυτή τη συμφωνία είναι λογική. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ε, υποχρεωτικές διατάξεις για τους γεωργούς περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επίσης, ε, οι γεωργοί που αναβαθμίζουν τα φιλοπεριβαλλοντικά τους ε, κριτήρια και πρότυπα συμβάλλουν στην υλοποίηση των ε, περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη και τα εθελοντικά μέτρα των γεωργών για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων είναι σημαντική συνεισφορά της γεωργίας στην Ευρώπη. Φυσικά θα πρέπει να παράγονται κυρίως υγιεινά τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους Γιώργους. Όχι η ποσότητα, ούκεν το πόλο το Φυσικά η ποσότητα θα πρέπει και αυτή να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ε, επάρκεια ε, διατροφική, γιατί έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά τα υγιεινά τρόφιμα είναι σημαντικό μας μέλημα και ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ευχαριστώ. Επερώτησε ο κύριος Τσόλος ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Τώρα στα πλαίσια της ίδιας ερώτησης αναφερθήκατε σε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν κατά της αρπαγής γεών. Ως προς αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω αν πιστεύετε ότι ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και μια τέτοια διάσταση, μια τέτοια διάσταση που να έχει να κάνει με τα αγροτεμάχια, με τα γεωργικά εδάφη, όσον αφορά τις διαπραγματεύσει που γίνονται στα πλαίσια της γεωργικής αγοράς. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να ακολουθούμε πάντα τους κοινοτικούς κανόνες, αλλά πολλές φορές υπάρχει και εθνική πτυχή, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τι επιλογέ που κάνει ένας γεωργός. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα οποιαδήποτε πολιτική ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί και την προσωπική επιλογή που ενδεχομένω να κάνουν κάποιοι γεωργοί προκειμένου να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένε αγροτικέ περιοχέ. Νομίζω ότι θα ήταν ε, θετικό να δείξουμε ότι ε, τα γεωργικά εδάφη αποτελούν πραγματικά ένα πολύτιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο. Σα ευχαριστώ. Αναμφίβολα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τσόλος. Είναι εθνικό, εθνικός σπόρος και η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι ευρωπαϊκός σπόρος. Δεν είναι ένα απλό προϊόν. Δεν είναι απλά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα. Είναι πραγματικά αγαθά και συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση σας. Και θα μπορούσαμε να συντάξουμε κάποια έκθεση για την πρόσβαση στην, ε, στις ευρωπαϊκές γεωργικές γης Γιατί όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Κούσμιουκ, είναι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες ε, που διέπουν την πρόσβαση των γεωργών στη γη. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν ευρωπαϊκό απολογισμό. Βέβαια τα θέματα κυριότητας των γεών είναι εθνική αρμοδιότητα και υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ των χωρών μελών, ιδιαίτερα χώρε χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Πάντως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διευκολύνουμε τους γεωργούς και την πρόσβασή τους στη γη. Ευχαριστώ. Κυρία Μόρτλερ, έχει τώρα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Οριστέντα Επίτροπε Βουιτσεχόφσκι. Στη Γερμανία κυριαρχεί το θέμα της βιωσιμότητας, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, όλο και περισσότερο σε αυτό το πλαίσιο ζητείτε 100% στροφή στην βιολογική γεωργία, στην οργανική γεωργία. Ποια είναι η άποψή σας, μπορούμε να έχουμε βιολογική ε, γεωργία, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για καλές και κακές ε, γεωργικές μετάσεις, καλούς και κακούς γεωργούς, τους βιολογικούς και άλλους. Ε, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, αν θέλετε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να γεφυρώσουμε τις δύο αυτές μορφές και η, φυτοπροστασία δεν είναι πιο βιώσιμη από την ε, έλλειψη παντελού, παντελή έλλειψη της φυτοπροστασίας. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως είπα, η βιολογική γεωργία είναι σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων τη κοινή γεωργικής πολιτικής και τη συμβολή της κοινή γεωργικής πολιτικής για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους. Και φυσικά ε, είναι μεγάλη και η ζήτηση της βιολογικής γεωργίας από τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και γι' αυτό έχουμε και ένα νέο κανονισμό για τη βιολογική γεωργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12,5 εκατομμύρια εκτάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούνται για βιολογική καλλιέργεια, βιολογική γεωργία και θέλουμε να αυξηθούν φυσικά αυτά τα εκτάρια. Και δεν είναι θέμα ε, διαμάχης ε, μεταξύ ε, βιολογικών γεωργών και συμβατικών γεωργών. Υπάρχει χώρος για όλους, αλλά η ζήτηση των καταναλωτών για περισσότερα βιολογικά προϊόντα έχει αυξηθεί και σίγουρα η βιολογική γεωργία θα πρέπει να ικανοποιήσει τι ανάγκε των καταναλωτών. Πάντως ε, η στήριξη τη ε, βιολογική γεωργία δεν γίνεται ει βάρο των συμβατικών γεωργών. Ούτε θέλουμε να εξαναγκάσουμε του γεωργού, να εγκαταλείψουν τη συμβατική γεωργία υπέρ τη βιολογική. Και οι παραδοσιακέ γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μερικές φορές είναι και εντατικής καλλιέργειας, χρειάζονται για να ε, υλοποιήσουμε την υπεσιτιστική μας ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια εναρμόνιση, γιατί και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε τη βιολογική γεωργία ε, για να ελοπίσουμε τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, χωρίς όμως να γίνεται αυτό εις βάρος της συμβατικής γεωργίας. Ευχαριστώ. Επερώτησα, σας ευχαριστώ. Κύριε Σαντε Επίτροπε, στις γραπτές σας απαντήσεις, αλλά και σήμερα μιλήσατε για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ε, για την ε, πρόθεση βουλική γεωργίας ε, και ότι θα καταθέσετε ένα τέτοιο σχέδιο. Το περιεχόμενό του μπορείτε να μας το πείτε. Τι θα κάνετε για την αγορά, τι θα κάνετε για τους καταναλωτές. Przepraszam, zdecydowanie e, Σίγουρα έτσι πρέπει να είναι το σχέδιο αυτό, όπως είπατε. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην γεωρική εκμετάλλευση. Άλλωστε αυτό προβλέπουν οι νομοθετικές διατάξεις. Αλλά αυτό είναι θέμα περισσότερο προώθησης ε, των βιολογικών τροφίμων και το θέμα της αξιοπιστίας του συστήματος θα πρέπει να γίνονται επαρκείς έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων, γιατί από μέχρι τώρα ελέγχους έχει προκύψει ε, πρόβλημα μερικές φορές σε τέτοια αξιοπιστία. Δεν είναι 100% σίγουρα αυτά τα βιολογικά προϊόντα, ότι είναι βιολογικά δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους ελέγχους και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των καταναλωτών σε σίγουρα και ασφαλή βιολογικά τρόφιμα, ώστε όταν ο καταναλώτης αγοράζει ένα βιολογικό γεωργικό προϊόν να είναι σίγουρος ότι πληρεί τις προσδοκίες του και τις, ανα... απαιτήσει του. Κυρία Πιντσέρνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε επίτροπε. Πριν από λίγο και σήμερα αλλά και στην προηγούμενη ακρόαση αναφερθήκατε στο Green Deal, στο ζήτημα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ξέρετε ότι τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και είναι ζητήματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ βέβαια και τους γεωργούς αλλά και τους καταναλωτές. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι το ακόλουθο. Θα μπορούσατε να μου πείτε πολύ συγκεκριμένα πώς θα καταφέρετε να πετύχετε τους δύο αυτούς στόχους. Και θα ήθελα και μία διευκρίνηση, διότι στις γραπτές απαντήσεις που δώσατε αναφέρεστε στην ε, επικουρικότητα και στις δυνατότητες που θα δοθούν στα κράτη-μέλη προκειμένου να καταφέρουν σε εθνικό επίπεδο να αντιμετωπίσουν και να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι ως προς αυτό χρειαζόμαστε μια εμβάθυνση, μια διευκρίνηση. Δεν πιστεύετε κύριε υποψήφιε επίτροπε ότι η δήλωσή σας αυτή ενδεχομένως να ερμηνευθεί ως κάτι το οποίο αντιβαίνει τελικά στην ίδια τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν η οποία είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει κεντρικό καθοριστικό ρόλο στον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δύο λεπτά, κυρία e, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, εγώ πιστεύω ότι οι προτάσεις για την κοινή γεωρική πολιτική που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα είναι πραγματικά μια επιθετική προσέγγιση. Πολλές υποχρεώσεις για τους γεωργούς. Βέβαια υπάρχουν και θετικές δράσεις που βελτιώνουν τη συνεισφορά της γεωργίας ε, στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Οπότε δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να αυξήσουμε αυτές τις ε, διατάξεις ή να τις κάνουμε πιο αυστηρές. Γιατί ήδη οι γεωργοί βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Τώρα αν εξαναγκαστούν σε δαπανηρές δράσεις που τους περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα θα βρεθούν σε ακόμη πιο δίνη κατάσταση. Ε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Και φυσικά αυτό το πράσινο οικοδόμημα που προτάθηκε και αυτή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ισορροπημένη μέχρι στιγμής γιατί επιτρέπει στο Γεωργό να συμβάλλει ενεργά στην ε, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τρόπο όμως ε, που θα τον ευνοεί. Γιατί μιλούμε για ισορροπημένη ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Ανάπτυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε, όταν μιλούμε για το μερίδιο των γεωργών και τη συνεισφορά τους στην, στο προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, θα πρέπει να αποβαίνει βάρος της ίδιας της γεωργίας. Γιατί Είπαμε ότι συμβάλλει η Γεωργία στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και την ίδια τη Γεωργία, γιατί αν εμφανιστεί τότε δεν θα έχουμε ούτε περιβάλλον ούτε κλίμα αν εξαφανιστεί η Γεωργία. Η προστασία της Γεωργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία και του περιβάλλοντος και του κλίματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τη συνεισφορά της γεωργίας σε αυτή την προστασία κλίματος και περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι δεν δώσατε όμως μια αρκετά διευκρινιστική απάντηση. Εσείς αναφερθήκατε στο ζήτημα της ευελιξίας. Ευελιξία που δίνεται στα κράτη-μέλη. Η ευελιξία αυτή δεν πιστεύετε ότι ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια διαδικασία επανεθνικοποίησης της κοινή γεωργικής πολιτικής που θέλουμε εμεί πάση θυσία να αποφύγουμε. Θεωρούμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λειτουργεί κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε από αυτού να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό έχετε Ευχαριστώ. Φυσικά υπάρχουν ε, αυτές οι ανησυχίες και οι φόβοι. Τους αντιλαμβάνομαι και μάλιστα τους εστερνίζομαι. Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολική επανεθνικοποίηση της Γεωργίας. Αλλά δεν συμφωνώ ότι η πρόταση του Επιτρόπου Χόγκαν για την νέα ΚΑΠ συνιστά ήδη επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Θα πρέπει πάντως ε, να δούμε αν αυτοί οι στόχοι χωρίς απαραίτητε κατευθυντήρε γραμμές εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και χωρίς συγκεκριμένους ε, δείκτε για την αξιολόγηση θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε του στόχους μας. Και επαναλαμβάνω, σε αυτή τη φάση θα διεξαχθεί η συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη φυσικά οι ανησυχίε σας και να διασκεδαστούν, γιατί αισθενίζομαι τους φόβους και τις ανησυχίες σα και στην πορεία της συζήτηση θα πρέπει να τους διασκεδάσουμε. Ευχαριστώ. Και προχωρούμε στο τελευταίο ερωτώντα, τον κύριο Μίχαλ Βίτσικ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο παραβλέψαμε στο πλαίσιο της ακρόασης αυτής η δασοκομεία. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κοινή ε, νοσιακή νομοθεσία όσον αφορά τα δασοκομεία. Υπάρχουν μόνο κάποιες οδηγίες που έχουν να κάνουν με, το, με τα ενδιαιτήματα και του οικότοπος. Ξέρετε ότι έχουμε την υλοτομία στην περιοχή Βιελοβίτζα στην Πολωνία που καταδεικνύει πραγματικά τη σημασία που μπορεί να έχει η κοινοτική νομοθεσία και είναι πάρα πολύ σημαντικές επίσης διαδικασίες επί παραβάση. Καθότι εσεί θα κληθείτε να ασχοληθείτε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα είπαμε για την βιοπικιλότητα θα πρέπει να ισχύουν και η δασοκομεία. Θα προωθήσετε εσεί μια τέτοια προσέγγιση. Επίση, ε, θα τηρήσετε μια τέτοια στάση ώστε να μην ανεχθείτε καμία παράβαση όσον αφορά την πολιτική δασοκομεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, Ευχαριστώ. Φυσικά και τα θέματα της δασοκομεία εμπίπτουν στι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική μέχρι στιγμής προστάτευε ε, τα ευρωπαϊκά δάση και τη δασοκομεία με πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και και στις ε, νέες προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπονται περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για τις έρευνες ε, για τα δάση. Και 182 εκατομμύρια εκτάρια δάση έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε στην κοινή γεωργική μας πολιτική να προστατεύσουμε και τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως διαφορετικά συστήματα και ίσως εκεί έγκυται το πρόβλημα στην πολύ διαφορετική κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη. Σε μερικά κράτη έχουμε ισχυρή δασική πολιτική, όπως στην Πολωνία, αναφέρατε το αρχαίγωνο δάσος Μπιγοβίτσα. Επίσης, άλλα κράτη χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των δασών. Αυτό είναι μια εθνική προσέγγιση. Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση, και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι το ελεκτικό συνέδριο ετοιμάζει μία έκθεση για την εφαρμογή και υλοποίηση αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δάση και τίποτα ουσιαστικά δεν θα αλλάξει, γιατί και στο παρελθόν στηρίζαμε στα δάση, στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να, να τα προστατεύουμε, γιατί είναι σημαντικός πλούτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δάση μας. Ευχαριστώ. Έχετε τώρα την επερώτησή σας. Ευχαριστώ. Αντιμετωπίζουμε δύο βασικές κρίσεις αυτή τη στιγμή. Κρίσεις που έχουν να κάνουν με την βιοπικιλότητα και κρίση που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις χρειαζόμαστε μία βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την βιώσιμη διαχείριση των δασών στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινή γεωργική πολιτικής. Ευχαριστώ. Λεπτό κύριε Φυσικά και υπάρχει σχετική υποστήριξη. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένη και βιώσιμη διαχείριση των δασών. Και αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δάση και θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής που επαναλαμβάνω ε, προτάθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται το 2013. Και ανάλογα με τον απολογισμό που θα κάνουμε και την αξιολόγηση, θα προγραμματίσουμε και θα σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα δάση. Πάντως, ε, δεν πιστεύω ότι η δασική πολιτική μας χρήζει αλλαγής είναι πολύ θετική. Βέβαια, έχουμε όλο και περισσότερες δασικές πυρκαγιές που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, οπότε έχουμε ένα επιπλέον επιχείρημα για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία του κλίματος και το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, γιατί τα δάση μας είναι πολύ ευάλωτα και είναι τα πρώτα θύματα των κλιματικών αλλαγών λόγω των αυξημένων δασικών πυρκαγιών. Οπότε, χρειαζόμαστε μία ε, πολιτική που θα προστατεύει το κλίμα και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Μάλιστα, αξιότιμοι συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Βοητσεχόφσκι για τη συμμετοχή του. Να ευχαριστήσω και τους 13 ερωτώντες, ερωτήσαντες. Και θέλω να σα ευχαριστήσω και εσά, ε, κύριε Βουλτσιεχόφσκι για το ότι ήσασταν πολύ πιο συγκεκριμένο ε, στις απαντήσεις σας σε σχέση με την προηγούμενη ακρόασή σας, ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σας δώσω τώρα το λόγο να κλείσετε με μια παρέμβαση που δεν θα πρέπει να υπερβεί τα πέντε λεπτά αλλά θέλω να σας πω ότι στη μία το μεσημέρι θα συνεδράσουν εκ νέου και κλεισμένα των θυρών οι συντονιστές ώστε να αξιολογήσουν ε, την ε, ε, σημερινή αυτή ακρόαση και έπειτα θα καταλήξουν στην άποψή τους για το κατά πόσον ο οριστής επίτροπος έχει τα δέοντα προσόντα ώστε να αποτελέσει μέλο σώματο των επιτρόπων και να αναλάβει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Κύριε και έχετε το λόγο για να κλείσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, τη δεύτερη συζήτηση που είχαμε. Είχαμε την ακρόαση την περασμένη εβδομάδα και σήμερα μου δώσατε την ευκαιρία για μια νέα ακρόαση και σας ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα μου στείλατε ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα ότι από τον Μελλοντικό Επίτροπο Γεωργίας περιμένετε όχι μόνο διαλλακτικότητα και ανοιχτό δεκτικό προς το διάλογο και μόνο λόγια, αλλά δικαίως περιμένετε αποφασιστικές δράσεις υπέρ της προστασίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι έτοιμος για αυτές τις δράσεις. Για τη Γεωργία, για την Ήπεθρο. Και η Γεωργία και η Ήπεθρος μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Και αν κάποιος φοβάται ότι δεν είμαι γεωργός, θα ήθελα να τον καθησυχάσω, γιατί ίσως αυτό το θεωρείτε ως αδύναμο σημείο της γεωργίας σας. Σας διαβεβαιώ ότι εγώ στην Ήπεθρο ανατράφηκα. Μεγάλωσα στην οικογενειακή αγροτική μας εκμετάλλευση και είδα πόσο σκληρή είναι η ζωή του Γιώργου, γιατί για πολλά χρόνια ασχολήθηκα με αυτό. Οπότε κατανοώ πλήρω τη γεωργική δραστηριότητα και είμαι πολύ ευαίσθητος απέναντι στα γεωργικά θέματα. Έχω αυτή την ευαισθησία λοιπόν, σας διαβεβαιώ. Και θα ήθελα ειλικρινά να δράσω υπέρ της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, υπέρ των γεωργών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και τα κατανοώ. Και φυσικά στο χρόνο μιας ακρόασης δεν μπορεί κανείς να απαντήσει διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις. Ακόμη δεν ε, είχα την ευκαιρία να κατατοπιστώ ε, δελεχώς για όλα τα θέματα, οπότε δεν μπορούσα να σας δώσω πολύ λεπτομεριακές απαντήσεις. Από τη στιγμή που γίνει κανείς επίτροπος θα εγκύψω όλα αυτά τα θέματα και θα ενημερωθεί πιο εμπεριστατωμένα. Και στα 12 χρόνια που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε συνεργασία μαζί σας, ενημερώθηκα για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και αξιώθηκα εξοικειώθηκα με αυτά. Καταλαβαίνω τη γεωργία και με την ευρωπαϊκή μου εμπειρία μπορώ να συμβάλλω σε μια ε, βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία και ανάπτυξη της ε, υπαίθρου, γιατί πραγματικά έχω αντιληφθεί πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή γεωργία. Και πιστεύω ότι χάρη στη συνεργασία που είχαμε και χάρη στη γνώση που έχω αποκομίσει, θα μπορέσω να δράσω για την ανάπτυξη της γεωργίας, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και να επιτελέσω το έργο μου προς το συμφέρον των γεωργών, αλλά και για το καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Περατούτε εδώ η συνεδρίαση και όπως είπα θα αρχίσει στη μία συνεδρίαση των συντονιστών.